Good afternoon, Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι έχουμε ε, παρκή ε, πλειοψηφία. Έχουμε παρτία για την σημερινή μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα το απόγευμα. Ξέρω ότι οι περισσότεροι είστε ιδιαίτερα απασχολημένοι σήμερα με τα διάφορα καθήκοντα. Έχουμε μόνο δύο σημεία στην ημερησία διάταξη, ψηφοφορίες και τα διάφορα αν δέχεστε την ημερήσια διάταξη, ε, να σα πω και ένα μήνυμα από του διερμηνεί. Βρισκόμαστε στην 21η μέρα των κινητοποιήσεων και ακόμα δεν έχουμε δει καμία αντίδραση εκ μέρου τη διοίκηση. Ο Γενικό Γραμματέα αντίθετα κληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση του. Στη σημερινή οι πολλοί συνάδελφοί μα από όλε τι καμπίνε έχουν επιταχθεί και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν σε ένδειξη λεγγύη. Η ελληνική καμπίνα δεν θα προχωρήσει σε στάση εργασία όπω αρχικά προβλεπόταν. Ωστόσο, η διερμηνία θα διακοπεί ακριβώ την προγραμματισμένη ώρα λήξη τη συνεδρίαση. Αυτό ήταν το μήνυμα από του διερμηνεί support them. Εμείς υποστηρίζουμε τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος, στο έργο τους. Ακούσατε το μήνυμα των διερμηνέων. I don't hear anything. Oh, that's it. Okay. Ωραία. Uh, thank you. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε με το πρώτο σημείο στην ημέρση διάταξη. Ψηφοφορία για μια έκθεση. Ο, κυρία, η κυρία Τόμα είναι η συγγήτρια, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήρθαν, γιατί κάποιοι ήρθαν μόνο για αυτή τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε εγκαίρω σε συμφωνία, έτσι ώστε τα κρατημένοι να μπορούν ε, να υποβάλουν έτσι για αυτό το πρόγραμμα που ξεκινά φέτο τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στην ψηφοφορία και να ξεκινήσουμε με την τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 και 37 και έμπλ 13 είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. η, καταπίπτει η έμπλ 12 γιατί απορρίφθηκε η προηγούμενη. Πάμε στην τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτονται. Τροπολογία 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Μπάτζετ 9 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία για την budget 9. The vote is closed. Λήξη. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο. Περνάμε. Εκόν 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Όχι. Είναι ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε στην τροπολογία 40 και έμπλη 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 41, Έμπλη 15, ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Έμπλη 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εκόν 1 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Εκον 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκον 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκον 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 4 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε. Έμπλ 4 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά για να δούμε. Λήξη. Απορρίπτεται. Λυπάμαι. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκόν 13. Καταπίπτει εμπλεφτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 4. Αποσύρεται 26, σωστά, ωραία. Πάμε στην τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. εποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. εποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην πλενιά, 9 υπέρ. Κατά. εποχές. Εγκρίνεται. Εκόν 15 υπέρ. Κατά. εποχές. Εγκρίνεται. Έμπλε 10 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τώρα να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στην κυρία Τόμασιτς. And we need to vote on... Και πρέπει να ψηφίσουμε για την εντολή για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is closed. Λήξη. Εγκρίνεται η εντολή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ψηφοφορία. Um, any other business for today? Υπάρχει κάτι στα διάφορα. Όχι, ευχαριστώ. Επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα, 9 Ιουλίου, το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνω τη συνεδρίασή μας.